Uh, Καλησπέρα σας. Συνεχίζουμε τη συνεδρίασή μας με τη συζήτηση των τροπολογιών του σχεδίου έκθεσης για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο Συντονισμού των Οικονομικών Πολιτικών και της εφαρμογής των προτεραιοτήτων για το 2013. Η συγκήτρια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό είναι η κυρία Φερέιρα. λέει Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά του εκπροσώπου των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ε, μας κάνουν μεγάλη τιμή με την παρουσία τους εδώ. Έχουμε διερμηνία από και προς 22 γλώσσες. Δεν θα εφαρμόσουμε το σύνθεση σύστημα του Catch the Eye. Δηλαδή να ζητά το λόγο ποιος τραβήξει την προσοχή του Προέδρου, αλλά θα δώσουμε πρώτα το λόγο στην κυρία Ελίζα Φερέιρα, την εισηγητριά μα, και μετά όποιο θέλει το λόγο, είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είτε από τα Εθνικά Κοινοβούλια, θα πρέπει να το δηλώσει στο φύλλο που θα κυκλοφορήσει, να το υποβάλει στους κλητήρες και οι κλητήρες θα το δώσουν στη γραμματεία. Ο κύριος Χέρμαν Τεκρό από την Βελγική Βουλή ζήτησε συγγνώμη για την απουσία του. Δυστυχώς ε, δεν θα παραστεί. Επαναλαμβάνω, αν θέλει κανείς το λόγο θα πρέπει να το δηλώσει στο φίλο που κυκλοφορεί. Συμπληρώστε το φίλο αυτό, δώστε το σε κάποιον κλητήρα και θα το ε, δώσει στη γραμματεία. και οι ευρωβουλευτές και οι σκιώδεις συγητές ε, θα πρέπει να ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία για να ζητήσουν το λόγο, να συμπληρώσουν δηλαδή αυτή τη σελίδα με τα στοιχεία τους και να τη δώσουν στον κλητήρα. Θα ήθελα να σας ενημερώσω και στους ευρωβουλευτές και στους εθνικούς βουλευτές ότι θα δίνω το λόγο εναλλακτικά σε δύο εθνικούς βουλευτές και έναν ευρωβουλευτή. Για κάθε δύο εθνικού βουλευτέ δηλαδή θα λαμβάνει το λόγο ένα ευρωβουλευτή. Ο χρόνο αγόρευση θα είναι τρία λεπτά το πολύ για τον κάθε ομιλητή. Σας θέρμο παρακαλώ να τηρήσετε αυτό το τρίλεπτο γιατί σίγουρα θα ζητήσουν πολύ το λόγο και έχουμε μόνο μέχρι τις 4.30 χρόνο για συζήτηση. Χωρίς άλλη καθυστέρηση θα δώσω το λόγο στη εισηγητριά μας, την κυρία Ελίζα Φερέιρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε κυρίως από τις Εθνικές Βουλές ε, στη συζήτηση αυτή. Μια συζήτηση που λαμβάνει χώρα ε, σε μια ιδιαίτερα επίκαιρη στιγμή. Αφενός γιατί ακόμη δεν έχουμε εξέλθει από την κρίση που έπληξε την Ευρωζώνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικώ τον κόσμο ολόκληρο. Πριν από πέντε χρόνια ακριβώς είχαμε την δόκευση της Lehman Brothers και η πτώση αυτή ε, έδειξε τα τροτά σημεία του ισχύοντος τότε μοντέλου. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι η ε, για ένα κείμενο που παρουσιάζει ένα νέο στοιχείο και που ευθυγραμμίζεται με την πρόσφατη έγκριση μιας ε, νέας μεθοδολογίας που ακολουθεί την ε, παράδοση του εξαπλού πακέτου και του διπλού πακέτου. Το εξαπλό πακέτο, το πακέτο των έκτο, έξι νομοθετικών προτάσεων ήδη έχει τεθεί σε ισχύ και αυτή τη στιγμή καλούμαστε να εξετάσουμε και να συζητήσουμε για μια πολύ σημαντική φάση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Έχουν ήδη γίνει οι συστάσεις ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Εγκρίνη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποβάλλει κάποιες τροπολογίες ε, στη διαδικασία αυτή της ε, λογοδοσίας. Ελπίζουμε ότι από το Ευρωπαϊκό αυτό εξάμεινο και από τις ε, συζητήσεις για τις ειδικές συστάσεις αναχώρα θα έχουμε μια καλύτερη συζήτηση για τα σχέδια προϋπολογισμών, εθνικών προϋπολογισμών και η συζήτηση αυτή θα γίνεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου λοιπόν περιμένουμε από τις χώρες μέλη στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου να υποβάλουν τα σχέδια προϋπολογισμού τους και οι ειδικές συστάσεις αναχώρα σχετίζονται με την πρώτη εκτίμηση που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτών των προσχεδίων προϋπολογισμού απότερο στόχος είναι να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή συνεργασία στα θέματα της διαχείρισης της οικονομικής πολιτικής. Έχω ήδη υποβάλει την έκθεσή μου, την έχω παρουσιάσει και από τις πολιτικές ομάδες έχουν υποβληθεί 230 τροπολογίες. Σε αυτή τη φάση προσπαθούμε να συμπεριλάβουμε στο μέτρο του δυνατού τις τροπολογίες στο κείμενο της έκθεσής μου με βάση την αρχή που ισχύει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια προσπάθεια δηλαδή ανέβρεσης ε, συμβιβαστικών λύσεων και όσο ευρύτερης δυνατή συνένεσης. Χάρη σε αυτή την προσπάθεια ελπίζω να καταλήξουμε σε ένα κείμενο που θα τύχει ευρείας αποδοχής χωρίς ε, αντίθετα να αλλοιώνονται οι βασικές ε, γραμμές, οι αδρές γραμμές του μηνύματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή τη δύσκολη φάση του ευρωπαϊκού βίου. Τώρα, ποια είναι τα διάφορα θέματα που περιλαμβάνω στην έκθεσή μου. Πρώτα απ' όλα προσπαθώ να δώσω μία όθηση στην πραγματική οικονομία. Θεωρώ ότι χωρίς αυτή την οικονομική ανάκαμψη δεν πρόκειται να ξεφύγουμε από την κρίση. Και στα πλαίσια αυτή τη οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη τεράστια αλληλεπίδραση που παρατηρείται μεταξύ των ε, ευρωπαϊκών οικονομιών, των οικονομιών των διαφόρων χωρών. Και η ευρωπαϊκή οικονομία δεν θα σταθεροποιηθεί αν προηγουμένω δεν γίνει ένα συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, ώστε να γεφυρωθούν αυτέ οι διαφορέ ανταγωνιστικότητε που παρατηρούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στην Ευρωζώνη χαιρετίζουμε κάποιες καινοτομίες που περιλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της και ιδιαίτερα το γεγονός ότι στην πρόταση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πρώτη φορά ασχολείται με σαφή τρόπο και αντιμετωπίζει με σαφή τρόπο την ανάγκη και τη σύσταση ακόμη και χώρες που έχουν πλεονάσματα να καταβάλουν προσπάθειες για να γεφυρωθούν αυτές οι ανισότητες και αποκλείς που υπάρχουν στην Ένωση. Βέβαια, οι χώρες αυτές που έχουν πλεονάσματα μπορούν να προωθήσουν την εσωτερική ζήτηση μειώνοντας ε, τα επίπεδα κοινωνικών εισφορών, διαπιστώνοντας ότι η εξέλιξη, η μισθολογική εξέλιξη τη χώρα αυτές θα πρέπει να συμβάλλει στην υλοποίηση του στόχου και ε, θα έχει θετικά αποτελέσματα και στην υπόλοιπη ευρωπαϊκή οικονομία. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε επανειλημμένως διαπιστώσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα λειτουργήσει εύρυθμα και αποτελεσματικά μόνο αν οι χώρες που έχουν πλεονάσματα και κάνουν προσαρμογές προσπαθήσουν να, να τονώσουν τη ζήτηση και υιοθετήσουν δυναμικές επενδύσεις. Αντίθετα, βραχυπρόθεσμα θα πρέπει να βρούμε κάποιες πολιτικές που θα καταπολεμήσουν την ανεργία, κυρίως την ανεργία των νέων. Και θα πρέπει να γίνουν και κάποιες σημαντικές μεταρρυθμίσεις και προσαρμογές ώστε να περιορίσουμε τους τεράστιους, τα τεράστια δυστυχώς ποσοστά φτώχεια και κοινωνικού αποκλεισμού. Χρειαζόμαστε λοιπόν και βραχυπρόθεσμε αλλά και μέσο και μακροπρόθεσμε πολιτικές για να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες και αποκλήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στην Ευρωζώνη και ταυτόχρονα να γνωρίσουμε ότι η ανταγωνιστικότητα φυσικά έχει κόστος αλλά χρειάζεται επενδύσεις, ανάπτυξη και διαπαιδαγώγηση και παιδεία προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα των κρατών μελών και ιδιαίτερα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ιδιαίτερα ε, είναι σημαντικό οι χώρες που έχουν έλλειμμα ανταγωνιστικότητας να εντείνουν τις προσπάθειές τους. Η έκθεση μου αναφέρει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναλύσουν τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο των μεταρρυθμίσεών τους και να γίνει μια αναθεώρηση των μοντέλων που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα. Γιατί διαπιστώσαμε και πολλά, πολλά και σοβαρά σφάλματα εκτίμησης των επιδράσεων και του αντικτύπου αυτών των πολιτικών. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό ιδιαίτερα για τις χώρες που θα πρέπει να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις γιατί για τις χώρες αυτές πολύ σημαντικά λάθη έχουν γίνει στις προβλέψεις και αυτό είναι δύσκολο να το εξηγήσουμε στους Ευρωπαίους πολίτες. γιατί υπήρχαν λάθη εκτιμήσεις και της πραγματικής οικονομίας και των μακροοικονομικών δικτών. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια συντονισμού στα πλαίσια της οικονομικής και νομισματικής μας πολιτικής, ταυτόχρονα να αξιοποιήσουμε τα κείμενα του εξαπλού πακέτου και να μειώσουμε τις μακροοικονομικές ε, ανισορροπίες και φυσικά να διεκπαιρεώσουμε τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έχουμε συμφωνήσει. Θα πρέπει όμως οι διαρθρωτικές αυτές μεταρρυθμίσεις να προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας και να γίνονται με την ελαστικότητα που προβλέπουν το εξαπλό και το διπλό νομοθετικό πακέτο και με τρόπο ανάλογο με τους στόχους που υλοποιούν, ώστε να μην έχουμε τον ολέθριο και η δραματικό αντίκτυπο που ουσιαστικά είναι αντίθετος από αυτο που αναμέναμε σε κοινωνικό επίπεδο. Αυτή η εξυγίαση οικονομική, δημοσιονομική λαμβάνει υπόψη φυσικά την αλληλεπίδραση των οικονομιών των διαφόρων χωρών μελών και φυσικά είναι και ένας ε, συναγερμός ε, ώστε να μην ξεχάσουμε τη μεγάλη σημασία που έχουν οι επενδύσεις. Γιατί χάρη σε αυτές ε, θα υλοποιήσουμε τους στόχους ε, τη στρατηγική του 2020 και θα φτάσουμε σε μια βιομηχανική πολιτική πραγματικά ευρωπαϊκή. Όλοι αυτοί οι επιμέρου τομεί λοιπόν θα πρέπει να επανεξεταστούν και δίνουμε κάποια στοιχεία στα κείμενα που έχουμε υποσυζήτηση. στοχο μα επαναλαμβάνω, είναι το συντομότερο δυνατόν να επιτύχουμε μια ανάκαψη τη οικονομια μια τόνωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μία αναχέτηση της δραματικής κατάστασης που διαπιστώνουμε στην ανεργία και κυρίως στην ανεργία των νέων. Σε ό,τι αφορά τις χρηματοπιστωτικές αγορές, φυσικά μας απασχολεί το γεγονός ότι η ροή πιστώσεων προς την πραγματική οικονομία σχεδόν έχει διακοπεί και θεωρούμε ότι το έργο που γίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχουμε εδώ πολλούς συναδέλφους που ασχολούνται με τα θέματα αυτά, όπως και υποφαινομένοι, την περασμένη εβδομάδα εγκρίναμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το, την ενιαία ευρωπαϊκή εποπτεία, οπότε θα έχουμε έναν ενιαίο επόπτη, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για τις χώρες Ευρωζώνης και για τις χώρες που προεδρικά θα εισέλθουν στο σύστημα αυτό και θα συνεργαστεί φυσικά η Κεντρική Τράπεζα με την Ευρωπαϊκή Αρχή των Τραπεζών και τους εθνικούς επόπτες για τις χώρες που βρίσκονται εκτός της Τραπεζικής Ένωσης. Σήμερα στην Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή είχαμε μία έντονη συζήτηση για τον ενιαίο μηχανισμό εκαθάριση εξυγίασης των τραπεζών και τα ταμεία και τα κονδύλια που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν από τον κλάδο και που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να επιτύχουμε μια εκαθάριση εξυγίαση που μαζί με το bail δηλαδή τον μηχανισμό διάσωσης με ίδιους πόρους, ώστε το κόστος της εκαθάρισης να μην το λαμβάνουν οι φορολογούμενοι, αλλά οι πιστωτές και οι μέτοχοι κατά κύριο λόγο της τράπεζας, πιστεύουμε ότι έτσι δημιουργούμε τα θεμέλια για τη σταθεροποίηση των τραπεζών, τη διασφάλιση των φορολογουμένων, την εγγύηση των καταθέσεων και την επαναφορά των τραπεζών στην υπηρεσία της πραγματικής οικονομίας. Γι' αυτό και ζητούμε να ενισχυθεί ο αγώνας για την καταπολέμηση της, φτω... της ε, φορολογικής ε, απάτης, φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής, των φορολογικών παραδείσων και άλλων ατασταλιών και ανομαλιών των χρηματοπιστωτικών αγορών. Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να πω ότι είναι σημαντικό να μην χάσουμε και το δημοκρατικό έλεγχο. Είναι μεγάλη η ευρωπαϊκή φιλοδοξία στη διαδικασία αυτή. Είμαστε υπέρ της προσπάθειας που γίνεται προκειμένου να διαμορφώσουμε έναν ευρύ οικονομικό χώρο, που θα είναι όμως και χώρος οικονομική δημοκρατίας. Ε, γι' αυτό χρειαζόμαστε μηχανισμούς διαφάνειας και μηχανισμούς ανάμειξης και των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών. Και φυσικά η δράση της Τρόικας ε, θα πρέπει επίσης να υπόκειται σε δημοκρατικό έλεγχο και να εντάσσεται στο, στην κανονική μέθοδο λειτουργίας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή με απόδοση ευθύνης, με λογοδοσία και με το κανονικό δημοκρατικό έλεγχο. Έχουμε πάντως κάποια, κάποιες ενδείξεις πρόοδου που δεν περνάνε απαρατήρητες. Για παράδειγμα, το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις συστάσεις ε, αναχώρα ή φετινές ανοίγουν μέτωπα που μέχρι στιγμής ε, ε, δεν ε, λαμβάνονταν υπόψη στη συζήτηση και υπάρχουν και άλλα σημεία πρόοδου που θα ήθελα να σας αναφέρω. Το πρώτο είναι μια δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έγινε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά από απαιτήσει και κλείσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πλαίσια του διπλού πακέτου ώστε η ανάλυση των εθνικών προϋπολογισμών για το 2014 να συνοδευτεί από προγράμματα ε, εξυγίασης, ε, τόνωσης ε, της ανάπτυξης, της απασχόλησης και στο προληπτικό σκέλος του πακέτου. Έχουμε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ιδρυθεί μια ομάδα εμπειρογνώμων υψηλού επίπεδου προκειμένου να λυθεί η δυνατότητα έκδοσης από κοινού κοινών ομολόγων από τα κράτη-μέλη γιατί το πρόβλημα των του δημόσιου χρέους δεν έχει επιληθεί, οπότε έχει ήδη ε, συστηθεί αυτή η ομάδα εμπειρογνωμών, όπως είχαμε ζητήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια του διπλού πακέτου. Και επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση για την δημιουργία ενός ενιαίου μηχανισμού εκαθάρισης εξυγείας των τραπεζών, ώστε να μην πληρώνουν τα σπασμένα των τραπεζών οι φορολογόμενοι, αλλά οι ίδιοι οι μέτοχοι, οι δανειστές και το ταμείο εκαθάρισης που θα χρηματοδοτείται από τον ίδιο τον τραπεζικό κλάδο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα. Περιμένω φυσικά με ανυπομονησία τα σχόλια και τις παρατηρήσεις των συναδέλφων. Έτσι θα διαμορφωθεί μια σαφή θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα λαμβάνει όμως υπόψη και τις ανησυχίες των Εθνικών Κοινοβουλίων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Σας ευχαριστούμε θερμά Ελίσσα. Περάμε τώρα στη συζήτηση Ξεκινούμε από τη Γαλλία, από τον κύριο Κριστόφ Καρές, που είναι μέλος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. Σας υπενθυμίζω το τρίλεπτο που δικαιούται ο κάθε αγορητής και σας να παρακαλώ εκ των προτέρων να το τηρήσετε. Κύριε Καρές, έχετε το λόγο για τρία λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μπορούσα και εγώ να αναφέρω εδώ πέρα κάποια πράγματα που γνωρίζω από δική μου εμπειρία. Ως εθνικοί βουλευτές, τουλάχιστον εγώ στη Γαλλία, ως εθνικός βουλευτής, μπορώ να πω ότι διένυσα αυτόν τον πρώτο πραγματικό χρόνο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, που πρόκειται βέβαια να συνεχιστεί με το νέο νομοσχέδιο για το νέο μας προπολογισμό και βέβαια η Επιτροπή μας θα πρέπει να γνωμοδοτήσει για αυτό το νέο νομοσχέδιο προπολογισμού. Γενικά πρέπει να πω ότι ε, ο διάλογος ήταν επικοδομητικός και είχαμε ουσιαστικά δύο ζητήματα τα οποία ανέκυψαν και από αυτόν θα ήθελα να επιμείνω. Το πρώτο ζήτημα, πάντα βέβαια από την οπτική γωνία της Γαλλίας, το πρώτο ζήτημα λοιπόν έχει να κάνει με τον ε, ρυθμό τον οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε όσον αφορά δηλαδή τις ε, αποφάσεις που λαμβάνονται για το δημοσιονομικό τομέα. Έγινε από αυτού μια συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είδαμε επίση ότι υπήρξε μια κάποια αναβολή όσον αφορά κάποιους στόχους. Θεωρώ πάντως ότι η συζήτηση αυτή εμπλέκει βέβαια και την κυβέρνηση της Γαλλίας και εμπλούτησε αστικά τις αποφάσεις της, αλλά και την ίδια την Επιτροπή, γιατί ο αρχικός ρυθμός, το αρχικό χρονοδιάγραμμα αποφάσεων ήταν πάρα πολύ απόλυτο και ουσιαστικά πάρα πολύ δύσκολο για μας. Και είχε μια πολύ σημαντική δρακόντια επίπτωση θα έλεγα όσον αφορά τις δραστηριότητές μας αλλά ακόμα και την ανάπτυξη της οικονομίας μας. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που βλέπω ότι η Επιτροπή εισάκουσε την, το δικό μας το αίτημα, το έλαβε υπόψη της και νομίζω ότι είχε γίνει και μια γενικότερη ανάλυση της κατάστασης, η, η ανάλυση δηλαδή από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο αναγνώρισε ότι ενδεχομένως να είχαν υποεκτιμήσει τις συνέπειες μιας πολύ σημαντικής δραστικής δημοσιονομικής προσαρμογής. Αυτό είναι το πρώτο ζήτημα το οποίο ήθελα να θίξω. Το δεύτερο τώρα ζήτημα έχει να κάνει με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Και πιο συγκεκριμένα, σε ποιο σημείο φτάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέχρι ποιο επίπεδο φτάνει στις συστάσεις της. Δηλαδή σε ποιο επίπεδο παρέμβασης φτάνει τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις εθνικές πολιτικές μέσω των συστάσεών της. Είναι σαφές ότι ως προς αυτό οι συστάσεις που γίνανε συγκεκριμένα προς τη Γαλλία για τις διαρθρωτικές μας μεταρρυθμίσεις ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένες και ουσιαστικά πηγαίνανε πάρα πολύ μακριά. Ουσιαστικά ήταν ε, πολύ ακραίες ή υπερβολικές οι συστάσεις. Προφανώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να θέσει μία σειρά από στόχους, από την άλλη όμως νομίζω ότι να στα κράτη-μέλη και στις εθνικές κυβερνήσεις και τα εθνικά κοινοβούλια στην πλειοψηφία δηλαδή που υπάρχει σε εθνικό επίπεδο να εφαρμόσουν τις αποφάσεις αυτές. Έτσι λοιπόν μια σχετική συζήτηση έλαβε χώρα στο Γαλλικό Κοινοβούλιο όταν είχε έρθει ο Επίτροπος Όλη Ρέ να μας μιλήσει Ήταν σαφώ επικοδομητική η συζήτηση αυτή, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να οριοθετήσουμε συγκεκριμένα τι αρμοδιότητε Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συγκεκριμένα προ τι συστάσει που απευθύνει προ τα κράτη-μέλη. Νομίζω το ζήτημα αυτό φάνηκε ξεκάθαρο όταν είχαμε αυτόν τον διάλογο μεταξύ Γαλλία και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε κύριε Καρέ. Εκ μέρου τη Ουγγρική τώρα Εθνική Βουλή, το λόγο έχει η κυρία Μαριά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Έγιναν ε, μεγάλες συζητήσεις σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες ε, συστάσεις, αλλά θέλουμε μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ της Κομισιόν και των κρατών μελών για να διευκρινιστεί η θέση του κάθε κράτους μέλους. Και αυτό θα πρέπει να γίνει γέρος βέβαια. Θα πρέπει οι συγκεκριμένες συστάσεις να χορηγούνται προς τα κρατη πιο νωρίς, προκειμένου να μην υπάρχει περιθώριο παρανόησης και θα πρέπει λοιπόν αυτό να γίνει προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση και θα πρέπει να ήταν πιο ευέλικτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά την τροποποίηση των συστάσεων και θα πρέπει να είναι και πιο ανοιχτή η στάση σε ό,τι αφορά τον πολιτικό κίνδυνο που ενέχεται στο καθεστώς της ιδιοκτησίας. Η Ουγγαρία ενδιαφέρεται ιδιαίτερως για το ευρωπαϊκό εξάμεινο και ο κύριος Ζωταντσίφικης έλαβε έλαβε οι πληροφορίες σχετικά με τις επόμενη προγραμματική περίοδο. Η Ουγγαρία δε δίνει ιδιαίτερη σημασία σε ό,τι αφορά τις συστάσεις, δαπανή κονδύλια για να βελτιώσει την κατάσταση. Θεωρούμε ότι οι μακρόπνοες μεταρρυθμίσεις και τα βασικά πολιτικά θέματα χρήζουν μεγαλύτερης προσοχής. Κατά την άποψή μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πάρα πολύ άκαμπτη σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες αναχώρας συστάσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις ε, μακροπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις. Ε, συμφωνώ με τον προηγούμενο μελετή. Συμφωνεί η Ουγγαρία με τις γενικότερες ε, προοπτικές και το γενικότερο προσανατολισμό των συστάσεων, αλλά θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη σημασία στο γενικότερο πλαίσιο, να δώσει μεγαλύτερο περιθώριο λιγμού στα κράτη-μέλη, σε ό,τι αφορά και τον τρόπο εφαρμογής των συστάσεων αυτών και τις λεπτομέρειες της εφαρμογής. Δεν είναι πάρα πολύ χρήσιμο, λοιπόν, να υπάρχουν αυτές τις συστάσεις αν ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τέτοιο ευρύ τρόπο ερμηνεύει τις αρμοδιότητές της. Σας ευχαριστούμε. Το λόγο έχει τώρα ο συντονιστής μας από το ΕΛΚ και σκιώδης συγγετής στην έκθεση κυρίας Φεραίρο, ο κύριος Γκοζές. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να τονίσω ότι ε, οι διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη με την εισηγήτρια και τους σκιώδεις ηγητές ε, λαμβάνουν χώρα σε ένα ιδιαίτερα θετικό και επικοδομητικό πνεύμα και είμαι σίγουρος θα καταφέρουμε να καταλήξουμε πολύ γρήγορα σε ένα πολύ θετικό συμβαστικό κείμενο όσον αφορά το σημαντικό και δύσκολο αυτό ζήτημα. Θα ήθελα να απαντήσω κάπως στις αντιδράσεις μόλις τώρα άκουσα για τις συστάσεις. Όταν ήμουν εισηγητής για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο στον πρώτο κύκλο, είχαμε συμφωνήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέγοντας ότι οι συστάσεις θα έπρεπε να ήταν λεπτομερείς. Και για ποιο λόγο λεπτομερείς για να καταφέρουμε να βγούμε από την ε, τυποποιημένη αυτή διατύπωση, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και μόνο αυτό, για να μπορούμε πραγματικά να αξιολογήσουμε την εφαρμογή των συστάσεων και πρέπει για αυτό το λόγο να έχουμε συγκεκριμένα κριτήρια, να ξέρουμε δηλαδή ποιοι είναι οι αρχικοί στόχοι που ετέθησαν και να είμαστε σε θέση να λάβουμε υπόψη μας και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και ως προς αυτό θα ήθελα να σας υπενθυμίσω κάτι πολύ σημαντικό. Ακούσαμε του συναδέλφου να μα μιλάνε για συστάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριο Μπαρόζο ενδεχομένω να έκανε κάποιο λάθο παρουσιάζοντα τι συστάσει αυτέ ω συστάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή τη στιγμή έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο. Οι συστάσει αυτέ δεν είναι πλέον συστάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι συστάσει που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι οποίε εγκρίνονται στη συνέχεια από τα κράτη-μέλη. Επομένω, οι συστάσει αυτέ είναι απόφαση των κρατών μελών. Επομένως είναι λανθασμένο να λέμε στη συνέχεια ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί αυτή τη στιγμή να επιβάλλει κάποιες αποφάσεις. Αν λαμβάνονται υπόψη και εφαρμόζονται συστάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι επειδή το επέτρεψαν και το αποφάσισαν τα κράτη-μέλη και μπορεί ένα κράτος μέλος να αποφασίσει κατά τη διάρκεια του εξαμήνου να αντιταχθεί στις συστάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να ζητήσει τροποποίησή τους οφείλουμε πραγματικά να αποσαφηνίσουμε το ζήτημα αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για να καταλάβει και ο Ευρωπαίος πολίτης πώς λειτουργεί το σύστημα. Αν δεν αποσαφηνίσουμε το σημείο αυτό, τότε θα αυξηθεί όλο και περισσότερο το χάσμα το οποίο υπάρχει μεταξύ Ευρώπης και Ευρωπαίων πολιτών. Και ξέρω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά να κατηγορούμε εύκολα την Ευρωπαϊκή Ένωση και προκειμένου την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι προκειμένου έχουμε συναπόφαση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτελεί αποφάσεις, αλλά η απόφαση λαμβάνεται από κοινού από του νομοθέτες Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να επενθυμίσω και κάτι ακόμα. Η εισηγήτριά μας μας προτείνει να κάνουμε μία εξάντε εις βάθος αξιολόγηση όλων των προτινόμενων μεταρρυθμίσεων. Συμφωνώ απόλυτα με την άποψη αυτή. Ωστόσο θεωρώ ότι θα πρέπει και να αναλύσουμε τι θα γινόταν αν δεν κάναμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Γιατί αν δεν υπήρχε ευρωπαϊκή ελληνική προς τις χώρες που βρίσκονται σε πιο δεινή κατάσταση, τότε οι χώρες αυτές θα βρισκόταν σε μια πολύ πιο δύσκολη κατάσταση από ό,τι βρίσκονται σήμερα. Επίσης, εγώ ουδέποτε πίστευα ότι η Ελλάδα θα έβγαινε από την Ευρωζώνη. Υπήρχαν και κάποιοι οικονομολόγοι οι οποίοι είχαν την ίδια άποψη, άλλοι πάλι που πίστευαν το αντίθετο. Βλέπουμε όμως σήμερα ότι χάρη στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά. Ξέρετε ότι ε, καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση χάρη στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και όχι μόνο χάρη στην διακυβερνητική μέθοδο. Χάρη στην αλληλεγγύη αυτή υπάρχουν κάποιες χώρε οι οποίε είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να προχωρήσουν προ μια κάποια ανάκαμψη. Αυτές τις παρεμβάσεις θέλω να κάνω, αυτή την παρέμβαση θέλω να κάνω και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποσαφηνίσουμε και να οριοθετήσουμε ακριβώς το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το ρόλο που αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη. Ας μην κατηγορούμε άδικα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τουλάχιστον για τα ζητήματα αυτά. Επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά ότι οι συστάσει αυτέ προτάθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά εγκρίθηκαν από τα κράτη-μέλη. Και ξέρω ότι χωρί τι συστάσει αυτέ δεν μπορούμε να έχουμε και τον ευκταίο συντονισμό των εθνικών πολιτικών. Σας ευχαριστούμε κύριε Γκοζές. Ήταν πολύ διαφωτιστική η παρέμβασή σας. Εκ μέρους του Κοινοβουλίου της Ιρλανδίας, το λόγο κύριος Λίντς, ο πρόεδρος της κοινή Επιτροπής Οικονομικών Δημοσίων Δαπανών και Μεταρρυθμίσεων. And... Σας ευχαριστώ πρόεδρε και εξ ονόματος του Ιρλανδικού Κοινοβουλίου θα θέλαμε να συμφωνήσουμε με τους ε, συναδέλφους και να ευχαριστήσουμε και εμείς με τη σειρά μας την κυρία Φεραίρα για την πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η έκθεση και για την πρόσκληση εδώ πέρα στην ε, Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Κύριε Πρόεδρε, όπως γνωρίζετε, από τον Σεπτέμβριο του 2010 συμμετείχε στο πρόγραμμα η Ιρλανδία και ε, επίσης 85 ε, δισεκατομμύρια ευρώ έχει λάβει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το EFSM, από τα, το EFSF, από το το, την ομάδα των χωρών που έχουν το ευρώ, από την Σουηδία, την Δανία και μέσω συμβολή της Ιρλανδίας μέσω του προγράμματος ε, συντάξεων. Όλα αυτά έχουν δημοσιευτεί σε σχέση με το πρόγραμμα αυτό. Στην παρούσα φάση η Ιρλανδία ε, επιτυχώς εφαρμόζει το πρόγραμμα, αλλά φυσικά θα πρέπει να σας πω ότι αυτό έχει γίνει εις βάρος των πολιτών που έχουν ε, υποστεί πολλές περικοπές σε ό,τι αφορά και τις δαπάνες τους. Σε ό,τι αφορά τον δημοσιονομικό έλεγχο, θα πρέπει να συγκεντρωθούμε και να επικεντρωθούμε στον τελικό απότερο στόχο, το να αποφέρει κέρδος απτό ε, η Ευρώπη εξερχόμενη από την κρίση κέρδος για τον πολίτη. Και σε κάποιες ε, ορισμένες αρκετές περιστάσεις ε, θέλουμε αυτό το μήνυμα να το μεταφέρουμε στον, στον πολίτη. Πώς λοιπόν μπορούμε να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη στην Ευρώπη, την ευημερία, την συνέχιση του κοινωνικού μοντέλου. Θα πρέπει να περάσουμε πέρα από τις ε, δαπάνες, τη, λιτότητα, να αρχίσουμε να μιλάμε και για ανάπτυξη, για ευημερία. Άρα συμφωνώ με την κυρία Φερέιρα και την έκθεση της ε, που καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγξει την ποιότητα της εφαρμογής όλων αυτών των μέτρων. Συμφωνώ επίσης ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις επενδύσεις και την αύξηση των επενδύσεων για την ανάκαμψη στην Ευρώπη. Και χαίρομαι που η κυρία Φερέιρα το ανέφερε αυτό και στην παρέμβασή τη. Επίση, θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο πτυχέ τη οικονομική διακυβέρνηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ό,τι αφορά τα κοινοβούλια. Καταρχά, σε ό,τι αφορά το οικοδόμημα Τη επισκόπησης της κοινοβουλευτικής αυτή την ε, σε αυτόν τον κρίσιμο κλάδο της πολιτικής. Ε, η ΕΚΟΝ αντιμετωπίζει το θέμα του προγράμματος για το 2013 και το 2014 και σύντομα θα, περάσουμε και θα πάμε και στο Vilnius που διοργανώνει λόγω της Λιθουανικής Προεδρίας σχετικό συνέδριο ε, το επόμενο έτος έχουμε και μια κοινοβουλευτική εβδομάδα που διοργανώνει η Προεδρία και το Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό. Άρα έχουμε τέσσερα συνέδρια σε τέσσερι μήνε. λίγο πολύ στα ίδια θέματα πολιτική. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξή. Τι θα έχουμε πετύχει ω τότε. Ποια θα είναι η αξία, ποιο θα είναι το κύρος που θα έχει το κάθε συνέδριο σε ό,τι αφορά το EGS. Μία ερώτηση λοιπόν έχω να ρωτήσω και το ρωτώ αυτό με ανοιχτό πνεύμα είναι αυτό ο αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπιση. Μήπω υπάρχει κάποιος καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό, γιατί θεωρώ ότι ίσω να υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη να ανταλλάσσουν απόψεις ε, οι βουλευτέ από τα εθνικά κοινοβούλια και έτσι νομίζω μπορούν να ασκήσουν καλύτερο έλεγχο στα εθνικά κοινοβούλια που τελικά, στις εθνικές κυβερνήσεις που τελικά παίρνουν τι αποφάσει στα κράτη-μέλη. Και θα έπρεπε λοιπόν ίσως να συζητούν ε, οι βουλευτές από τα Εθνικά Κοινοβούλια και από το Ευρωκοινοβούλιο πιο ευρεία θέματα. Δεν ξέρω κατά πόσον η διοργάνωση και το πρόγραμμα των συνεδρίων ε, εξυπηρετούν τους σκοπούς και του Ευρωπαϊκού και των Εθνικών Κοινοβουλίων σε ό,τι αφορά τα προπαρασκευτικά αυτά ε, έγγραφα. Δεν είμαι βεβαίως ότι αυτά εξυπηρετούν το σκοπό μας. Πώς θεωρείτε ότι θα πρέπει λοιπόν να δούμε αυτή τη σχέση μεταξύ αυτών των συνεδρίων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λέει και ο Πρόεδρος κύριε Λίντς. Και τώρα το λόγο έχει... Να δώσω το λόγο τώρα στον Πρόεδρο ε, της Επιτροπής Οικονομίας ε, από την Ισπανική Βουλή. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε, κύριο Σλανθουέλα. Χαίρομαι ιδιαίτερος ε, που ξαναβρίσκω τους συναδέλφους από τις ε, βουλές των χωρών μελών. Έχουν περάσει 13 μήνες που το spread ε, της Ισπανίας ξεπερνούσε τα, τις 600 μονάδες βάσης. Σήμερα το πρωί το spread ε, έφτασε στα 244. Μέσα 13 μήνες περάσαμε, μέσα σε 13 μήνες περάσαμε από 600 και βασικές μονάδες σε 244. Αυτό σημαίνει πολλά. Καταρχήν, ε, σημαίνει ότι η κυβέρνησή μας ακολούθησε πιστά τις συστάσεις της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και προέβη σε μία άρδιν ε, μεταρρύθμιση της οικονομικής πολιτικής στους τελευταίους 20 μήνες. Και συνεχίζεται αυτή η τεράστια οικονομική μεταρρύθμιση. Χρειάστηκε να γίνουν σημαντικές διορθώσεις των μακροοικονομικών ανισορροπιών που παρουσίαζε η Ισπανία πριν από μόλις 20 μήνες. Θα αναφερθώ σε τρεις τομείς. Καταρχήν έγινε η δημοσιονομική εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών, των δημόσιων λογαριασμών, κάτι που ήταν αναπόφευκτο για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των δημοσιονομικών της Ισπανίας. Επίσης, ολοκληρώθηκε μία ανακεφα... ανακεφαλαιοποίηση και αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα. Κάτι που διασκέδασε τις αφιβολίες για τη φερικιότητα του ισπανικού τραπεζικού τομέα. Και αναφίβολα, η εξυγίανση αυτή θα βοηθήσει στην ανάκαμψη της, της ροής των πιστώσεων και προς επιχειρήσεις και προς νοικοκυριά. Επίσης ε, έγιναν πολλές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην Ισπανία προκειμένου να ε, ανακάμψει η ανταγωνιστικότητά μας και η παραγωγικότητά μας. Και ήταν θεαματική και η αλλαγή στο εμπορικό μας ισοζύγιο μετά από τα μέτρα αυτά. Και επίσης ε, στο ισοζύγιο πληρωμών μας ήταν πολύ εντυπωσιακή η αλλαγή. Φυσικά θα συνεχίσουμε εφαρμόζοντας τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, γιατί όπως ανασωστά αναφέρθηκε δεν είναι οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά προτάσεις ολόκληρης ε, της Επιτροπής, λέει ο Πρόεδρος, ε, ο κ. Λασουέλα. Και σημαντικό είναι να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε αυτή την τεράστια πρόκληση που είναι η υλοποίηση μιας γνήσιας οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Και θέλουμε να συνεργαστούμε σε αυτή την προσπάθεια και σίγουρα η Φορολογική Ένωση και η Τραπεζική Ένωση θα είναι δύο τεράστιες προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως έχουμε εμπιστοσύνη ότι με συνεργασία όλων μας θα καταφέρουμε και πρόθεσμα να υλοποιήσουμε αυτούς τους στόχους. Σας ευχαριστούμε κύριε Λανθουέλα. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Φιλίπ Ντεμπάκερ που είναι σκιώδης ηγητής των Φιλελευθέρων. Eh, Ευχαριστώ Πρόεδρε και θα ήθελα καταρχάς ε, να καλωσορίσω και όλα τα εθνικά κοινοβούλια για τον πολύ σημαντικό αυτό διάλογο τον οποίο διεξάγουμε σήμερα και να ξεκινήσουμε με αυτό που είπε και μόλις ο κ. Γκοζές. Πολύ σημαντικό. Στο τέλος κάθε διαδρομής ε, τελικά το θέμα είναι το πώς όλοι μαζί θα πετύχουμε και από την ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και από τα εθνικά θεσμικά όργανα να πετύχουμε την έξοδο από την κρίση και με ποιον τρόπο μπορούμε το θέμα της ιδιοκτησία ε, για τα μέτρα αυτά τα οποία πρέπει να αναλάβουμε, πώς μπορούμε να το ενισχύσουμε λοιπόν αυτό το θέμα της ιδιοκτησίας και πώς μπορούμε να πετύχουμε την ε, δημοκρατική νομιμοποίηση. Να επικεντρωθώ λοιπόν σε αυτά τα δύο πράγματα. Καταρχάς την ανάκαμψη, την επιστροφή σε μια φυσιολογική κατάσταση. Νομίζω ότι έχουν γίνει μεγάλα βήματα και μέσω της ε, ευρωπαϊκής καθοδήγησης σε ό,τι αφορά την δημοσιονομική πειθαρχία που δέχτηκαν τα κρατημέλη, αλλά και με τα βήματα που έχουν γίνει για τον καλύτερο έλεγχο των τραπεζών σε ό,τι αφορά την φυσιολογική τους λειτουργία χωρίς υπερβολικούς κινδύνους. Αυτά λοιπόν γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε συνεργασία με τα κρατημέλη. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά. Νομίζω ότι έχουν γίνει βήματα τα οποία ήταν πραγματικά, θα φανέντουσαν αδύνατα σε κάθε πολιτικό πριν από πέντε χρόνια. Ένα δεύτερο στοιχείο, σύμφωνα επίσης με τον κύριο Κοζές και αυτά που είπε πριν από λίγο, σε ό,τι αφορά το ownership, ε, την ιδιοκτησία, αν θέλετε, κάποιων συστάσεων που γίνεται για θέματα δημοσιονομικού Δημοσιονομική εποπτεία, ε, αλλά και τι συστάσεις που, που έχει εγκρίνει το Συμβούλιο. Και φαίνεται λοιπόν ότι συνεχίζεται από τη συζήτηση που προκύπτει από τα εθνικά κοινοβούλια, ότι συνεχίζεται η αμφισβήτηση, αν θέλετε, η συζήτηση για τα θέματα αυτά. Παρά το γεγονός ότι πιο πολύ πλήττονται τα εθνικά κοινοβούλια από ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα λέτε ότι παίρνουν αποφάσεις. Όχι, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι αυτό που παίρνει αποφάσεις και που αυτό υποχρεούται μετά να εκπληρώσει τις αποφάσεις που λαμβάνει. Είναι λοιπόν σημαντικό να ξέρουμε μεταξύ σκύλας και χάριβδης σε ό,τι αφορά τις υπερβολικές δαπάνες, σε ό,τι αφορά την αναδιάθρωση και τις διευθυντικές μεταρρυθμίσεις, το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία αποφασίζουν αυτό από εμά ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τι, τι προαπαιτεί μια δέσμευση σε ό,τι αφορά την δική μας υποχρέωση, αλλά θεωρώ ότι και από τα Εθνικά Κοινοβούλια προαπαιτεί μια πιο έντονη συζήτηση με τις εθνικές κυβερνήσεις για την τοποθέτησή τους στο Συμβούλιο σε ό,τι αφορά τα μέτρα αυτά για την οικονομική ανάκαμψη. Και κλείνοντας πρόεδρε να πω το εξή. Νομίζω ότι οι συστάσεις, οι συγκεκριμένες αναχώρα είναι πιο πολύ από ποτέ απαραίτητες αν θέλουμε να επανέλθουμε σε ένα είδους φυσιολογική λειτουργία. Όπως είπε και η κυρία Φερέιρα, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υπάρχει κάποια σύγκληση αφενός μέσω του ελέγχου και της εφαρμογής των διαφορετικών μεταρρυθμίσεων και μάλιστα με πολύ λεπτομερή τρόπο όπως συμβαίνει σήμερα και κατά δεύτερον σε ευρωπαϊκό επίπεδο να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη στις επενδύσεις τους σε ό,τι αφορά σε υποδομές, σε καινοτομία, έρευνα. Θεωρώ ότι αυτά είναι κρίσιμη σημασία στοιχεία για την επαναφορά της ε, φυσιολογικότητας, αν θέλετε, και καλωσορίζω αυτή τη σημερινή συζήτηση με απότερο σκοπό να επανέλθουμε σε μια κανονική κατάσταση, να εξέλθουμε από την κρίση προς όφελος του πολίτη πάντα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Τεμπάκερ. Εκ μέρους της ε, ε, Εθνικής Βουλής της Σλοβενίας, το λόγο κύριο Φρέγκε, που είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής ε, Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων της Σλοβενικής Βουλής. Τρία λεπτά, μην ξεχνάτε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω με κάποιες κριτικές. Ε, λέμε ότι ο διάλογο αυτό είναι σημαντικός. Συμφωνώ. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια και μιλάμε για μακροοικονομική διακυβέρνηση. Δεν θα πρέπει όμως να ξεχνούμε ότι αφιερώνουμε μόλις μια μισή ώρα για το θέμα αυτό. Μα τι να προλάβει κανείς σε μια μισή ώρα. Πώς μπορούμε να μιλήσουμε με λεπτομέρειες για κάθε χώρα μέλη. Μέλος. Και ταυτόχρονα μιλούμε για τις ευρωπαϊκές συνέπειες ε, μιας τέτοιας συνεργασίας και ενός τέτοιου διαλόγου. Χρειαζόμαστε φυσικά αυτό το διάλογο και έχουν πολλές απορίες στα εθνικά κοινοβούλια και η πιο σημαντική απορία είναι το κατά πόσο οι συστάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανταποκρίνονται στην ιδιαιτερότητα της κάθε χώρας. Πολύ φοβάμαι ότι δεν είναι θέμα αν είμαστε ικανοποιημένοι, δυσαρεστημένοι με τις ε, συστάσεις, αλλά φαίνεται ότι είναι για μας το τελεσμένο γεγονός αυτές οι συστάσεις, ιδιαίτερα για την πατρίδα μου ε, που αυτή τη στιγμή έχει τη φήμη ότι είναι η επόμενη στη σειρά. Αν και η κρίση στη Σλοβενία είναι διαφορετική και η κρίση στον τραπεζικό τομέα και η υπερχρέωση της οικονομίας δεν σημαίνει ότι θα είναι η Σλοβενία η επόμενη στη σειρά της διάσωσης ο καλύτερος τρόπος ε, για την εξυγίαση των ε, δημοσίων οικονομικών είναι η τόνωση της ε, οικονομικής μεγέθυνσης. Θα πρέπει λοιπόν να διαρωτηθούμε κατά πόσο το ισχύον μοντέλο πραγματικά δημιουργεί δυνατότητες για ανάπτυξη και θέσεις απασχόληση, μήπως αντίθετα αναχαιτίζει την υλοποίηση αυτών των στόχων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις συστάσεις, οφείλω να ομολογήσω ότι τα κοινοτικά θεσμικά όργανα δεν ε, μας είπαν τίποτα καινούριο, τίποτα που δεν γνωρίζαμε ήδη στη Σλοβενία. Αυτό ισχύει ε, και για την τραπεζική κρίση και για την υπερχρέωση της οικονομίας. Αυτά τα γνωρίζαμε, δεν χρειαζόταν μας τα από τα θεσμικά όργανα. Και πέρσι και φέτος παρόλα αυτά η Σλοβενία ευλαβικά εφάρμοσε τις συστάσεις και μάλιστα βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο της ε, προετοιμασίας του προϋπολογισμού για το επόμενο έτος. Αλλά ήδη δημιουργείται μια κοινωνική διαμαρτυρία εξαιτίας αυτής της διαδικασίας. Σε ό,τι αφορά τις εκθέσεις, θα ήθελα να πω ότι έχουμε πολλές ιδιαιτερότητες και ίσως διαφορετικές ευαισθησίες ε, μεταξύ κοινού και κοινοβουλίου. Αυτό όμως ε, εντείνει την ευθύνη μας για τους επόμενους μήνες, γιατί θα πρέπει ως Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδείξουμε ότι είμαστε ικανοί να αντιμετωπίσουμε αυτή την οικονομική και κοινωνική κρίση. Πριν δεχθούμε την ψυχρολουσία α, της ανόδου των ευρωσκεπτικιστών στις ευρωεκλογέ. Είναι σημαντικό λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν ε, θα έρθει από μόνη της. Στην Αθηνά και χειρακίνη. Θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες ε, και να θέσουμε σε πράξη τα ωραία λόγια που λέμε. Σας ευχαριστώ κύριε Φέρεφ. Εκ μέρους της Λετωνίας τώρα, το λόγο κύριος Οσόλινς, ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών. Uh, thank you, sir. Uh, Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Το Εθνικό Κοινοβούλιο της χώρας μου συμμετέχει έντονα στο διάλογο όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και την ε, εφαρμογή των ε, ειδικών αναχώρα συστάσεων. Στα τέλη Μαΐου του 2013 ειδικέ αναχώρα συστάσεις παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή μας, την αρμόδια Επιτροπή του Κοινοβουλίου μας και Υπήρχε μάλιστα και επίσκεψη του Πεκεφαλή Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη συνέχεια, ο Υπουργό Οικονομικών μα ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την διαδικασία εφαρμογή των συστάσεων αυτών. Όσον αφορά τώρα την ε, εθνική κυριότητα των συστάσεων αυτών, πιστεύω ότι μπορεί να αυξηθεί η κυριότητα αυτή, ιδίως όσον αφορά την υποβολή των ε, σχεδίων συστάσεων. Θα θέλαμε να μπορούσαμε να λαμβάνουμε τις στάσεις αυτές κάποιες μέρες νωρίτερα, ώστε να μας δίδει το απαραίτητο χρόνος για να κάνουμε μια εισβάθος ανάλυση και να μην απαντάμε μόνο με ένα ναι ή με ένα όχι. Ιδίως όταν τα όσα προτείνονται έχουν να κάνουν με μακροπρόθεσμα προγράμματα προσαρμογής όταν χρειάζεται να μεταρρυθμίσουμε το σύστημα κοινωνική πρόνοιας ή το συνταξιοδομικό μα σύστημα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό απαιτεί πάνω από δύο-τρει μέρε όσον αφορά την συζήτηση σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Τώρα επανέρχομαι στις ειδικέ αναχώρα συστάσεις. Κάθε φορά που συζητάμε την χρηματοδότηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και όσον αφορά τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν σε εθνικό επίπεδο, εμείς θεωρούμε ότι όσα προβλέπουν είναι σωστά και ότι δεν θα οδηγήσουν σε δευτερογενείς επιπτώσεις. Επομένω δεν θέτουμε να αμφιβόλω τα όσα λέγονται. Όσον αφορά την δημοσιονομιακή πειθαρχία, προσπαθούμε να αντλήσουμε τα διδάγματα του παρελθόντος και ουσιαστικά συνειδητοποιούμε ότι μια αυστηρή δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να είναι ακρογωνιαίος λίθος μιας οικονομικής πολιτικής που θα ακολουθήσει η χώρα μου. Και αυτή τη στιγμή εγκρίνουμε, μάλλον στις αρχές του 2013 εγκρίναμε μια νέα νομοθεσία δημοσιονομικής πειθαρχίας, πραγματικά πρόκειται να αλλάξει εντελώς την ε, εκτέλεση της δημοσιονομικής πολιτικής ε, στην χώρα μου και θα οδηγήσει ουσιαστικά σε μια μακροοικονομική σταθερότητα και θα μειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις από εξωτερικούς παράγοντες που πειράζουν την οικονομία μας. Όσον αφορά την ενδυνάμωση του πλαισίου δημοσιονομικής πολιτικής, θεωρούμε ότι χρειαζόμαστε την απαραίτητη χρηματοδότηση για ένα νέο συμβούλιο χρηματοοικονομικό, το οποίο θα αρχίσει να λειτουργεί από το 2014 και που θα έχει ως στόχο να επιβλέπει την εφαρμογή των αποφάσεων στα πλαίσια της νομοθεσίας δημοσιονομικής πειθαρχίας. Το συμβούλιο αυτό θα απαρτίζεται από 3 με 6 ρετά μέλη. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσετε το λόγο και προσβλέπω σε περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων. Σας ευχαριστούμε κύριε Όζολης. Εκ μέρους των συντηρητικών δώρα και μεταρρυθμιστών, το λόγο έχει ο Σέπινγκ που είναι και σκιώδης ηγητής. Ε, Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα, γιατί πολλά ακούσαμε, να αναφερθώ σε αυτά που είπε ο κύριος Κάβες από τη Γαλλία. Ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό που έθιξε. Τι θα μείνει, τι θα απομείνει σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των Εθνικών Κοινοβουλίων, αν τα συγκρίνουμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε ό,τι αφορά την ροή των αρμοδιοτήτων που έρχεται προς τις Βρυξέλλες. Εγώ είμαι υπέρ του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που πρότεινε η κυρία Φερέιρα. Βλέπουμε ότι η Ευρωζώνη είναι ε, θέλουμε να γίνει ένας ε, δημοσιονομικός, ε, μια δημοσιονομική ένωση με κάποιες συστάσεις αναχώρα. Αναφέρεται ότι είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι υπάρχει εποπτεία για να ξέρουμε ότι πάει λάθος και ότι πρέπει να βελτιωθεί. Και έτσι καταλήγουμε στο ερώτημα ποια είναι η αρμοδιότητα του Εθνικού Κοινοβουλίου τελικά γιατί σε αυτή τη δημοσιονομική ένωση τα δημοσιονομικά δικαιώματα των εθνικών κοινοβουλίων, που είναι πάρα πολύ σημαντικά, ουσιαστικά παρακάμπτονται. Γιατί ο προπολογισμό γίνεται στις ε, Βρυξέλλες, περιορίζονται τα δικαιώματα των εθνικών κοινοβουλίων. Και έτσι δημιουργούνται ανισορροπίες. Τι σημαίνουν, τι σημαίνει αυτή η λέξη ανισορροπίες στον τραπεζικό τομέα στην Κύπρο. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ανισορροπίες για την Ιρλανδία, για τον κλάδο των ακινήτων στην Ισπανία, στην Ισπανία, στην ε, Ολλανδία, στην ε, Γερμανία έχουμε πλεονάσματα εμπορικά, στην Γαλλία, στην ε, Γερμανία μήπως η μισθή είναι πολύ χαμηλή, όπως είπε και ο Ευρωπαίος Επιτροπός για την Κοινωνική Πολιτική πρόσφατα. Αυτό φυσικά έχει να κάνει με κάθε εθνική πολιτική, κοινωνική, οικονομική στα κράτη-μέλη. Τι παραμένει λοιπόν μετά, τι θα απομείνει από τις δικές σας αρμοδιότητες. Κάποιοι προσπαθούν να πάνε και λίγο παραπέρα με οικονομικό συντονισμό εξάντε όπου ουσιαστικά κάθε πρόταση κάθε κυβέρνησης στον τομέα της οικονομικής κοινωνικής πολιτικής, για παράδειγμα, ή αναθεώρηση των ε, συντάξεων. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει πρώτα να υποβάλλονται στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες. Αυτό σημαίνει ότι ως συνομοθέτες οι αρμοδιότητές σας στο έτοιμο το κράτος μέλος σας θα περιοριστούν πολύ σημαντικά. Θα υποσκαφθούν ουσιαστικά περαιτέρω τα εθνικά κοινοβούλια. Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν την ισορροπία μεταξύ αυτού που η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει η Κομισιόν, το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο και αυτού που θα πρέπει να παραμείνει στα, χέρι, στα χέρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά, φυσικά το εκλογικό σας κοινό εσάς πρώτα θα κοιτάξει και θα πει τι κάνει το δικό μας το Κοινοβούλιο, η δική μας η Βουλή. Δεν προασπίζονται τα δικαιώματά μας. Αν λοιπόν οι εκλογείς δεν ε, καταλαβαίνουν τι έχει γίνει, πρώτα με εσάς θα θυμώσουν και πολύ μετά με εμά. Τίθεται λοιπόν θέμα νομιμοποίησης του συστήματος αυτού. Δεν αποτέχονται, ξέρετε, όλοι οι πολίτες να αποφασίζεται από, τις Βρυξέλλες η διαμόρφωση, για παράδειγμα, των ασφαλίσεων, των συντάξεων. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε μια λεπτή ισορροπία σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες των Εθνικών Κοινοβουλίων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των κρατών μελών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δούμε μήπως κάποια πράγματα θα πρέπει να παραμείνουν στα χέρια των κρατών μελών. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίνγκ. Εκ μέρους ε, της Πορτογαλικής Βουλής τώρα έχει το λόγο ο κύριος Κάπιτα που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής ε, Οικονομικών ε, και Δημοσιονομικών Θεμάτων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θεωρούμε ότι είναι σημαντική διεξαγωγή αυτής της συζήτησης γιατί μας επιτρέπει να κάνουμε μια πολιτική αξιολόγηση και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων μια πολιτική αξιολόγηση των ε, συστάσεων αναχώρα που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάρα πολλά όμως συμφωνούμε με το περιεχόμενο της έκθεσης κυρίας Φερέιρα που μας λέει ότι είναι απαραίτητο να δούμε πώς θα ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις που μας δημιούργησε η κρίση, ε, η οικονομική και η δημοσιονομική κρίση. Τη εβδομάδα αυτή που συμπληρώνουμε πέντε χρόνια μετά την πτώχευση της Lehman Brothers. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα διέλθουμε από την κρίση και την απάντηση στην, ε, στην πρόκληση της κρίσης θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε πανευρωπαϊκά και με ένα συντονισμό των πολιτικών μας, όχι μόνο βραχυπρόθεσμα, αλλά και μακροπρόθεσμα, προκειμένου να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για μια αηφόρο ανάπτυξη με δημιουργία θέσεων απασχόλησης και μέσο και μακροπρόθεσμα. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν η Πορτογαλική Βουλή συμμετέχει με ιδιαίτερο ενθουσιασμό στη συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο γιατί έχουμε επίγνωση ε, των ε, ειδικών προκλήσεων αυτής της ε, συζήτησης, ιδιαίτερα σε μια χώρα που βρίσκεται σε ένα πρόγραμμα διάσωσης και προσαρμογής που έχει συμφωνήσει με τους διεθνείς δανειστές της και ε, συμφωνώ με την εκτίμηση του Σλοβαίνου συναδέλφου ότι μια μισή ώρα είναι πολύ λίγος χρόνος για να συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Εμείς στην Πορτογαλική Βουλή προσκαλέσαμε την ε, κυρία Φερέρα για να μας παρουσιάσει την έκθεση την έκθεσή της ε, κατά την έναρξη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και ακούσαμε και την πρόεδρο της Επιτροπής την κυρία Σαρομβόλ που ήρθε στην Πορτογαλία και είχε συζήτηση με τους Πορτογάλους βουλευτές. Είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε μηχανισμούς τακτικής ε, συζήτησης και συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων και να μην ε, εξαρτώμαστε από κάποιες ε, περιπτωσιολογικές ή μεμονωμένες πρωτοβουλίες είτε του Κοινοβουλίου του Ευρωπαϊκού είτε των Εθνικών Βουλών. Πολύ πιστεύουμε ότι το ευρώ σώθηκε. Έχουμε ξεπεράσει το μεγαλύτερο τμήμα της κρίσης, αλλά κάποιος που είναι τόσο αισιόδοξο ε, ξεχνάει τις αιτίες της κρίσης, τις ανισορροπίες των χρηματοπιστωτικών αγορών που δημιούργησαν ασύμμετρα αποτελέσματα στις εθνικές οικονομίες και ξεχνάει τις, κοινωνικές αιτίε κάποιων ανελαστικών μορφών προσαρμογής που εφαρμόστηκαν. Η Πορτογαλία έκανε τεράστιες προσπάθειες για να τηρήσει τους εξωτερικούς της στόχους και υποσχέσεις. Αλλά με τις συστάσεις, όταν έχουμε αύξηση της ενεργείας, είναι δύσκολο να τις ε, τηρήσουμε. Πολλό δε μάλλον που βρισκόμαστε ήδη στο τέταρτο έτος της ύφεση. Γι' αυτό και θα πρέπει να ενισχύσουμε τον ευρωπαϊκό συντονισμό. Το διπλό πακέτο βαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Δεν θα πρέπει να σταματήσουμε τώρα να, συγκεκριμε... να συγκεκριμενοποιήσουμε την Τραπεζική Ένωση, συγκεκριμένους μηχανισμούς φορολογικής σύγκλησης, να ενισχύσουμε την ιδέα μιας γνήσιας οικονομικής και νομισματικής ένωσης στην Ευρωζώνη και στην Ευρώπη των 28 χωρών μελών και να μην ε, ε, βλέπουμε την κρίση σαν κάτι που δεν είναι ευρωπαϊκό αλλά κάτι που είναι ευθύνη η πετιότητα της α ή β χώρας. Για, την, για να ανταπεξέλθουμε στην κρίση χρειαζόμαστε μια κοινή απάντηση και αντίδραση. Σας ευχαριστούμε κύριε Καβρίτα. Τώρα εκ μέρους Σλοβενίας έχει το λόγο η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων, η κυρία Όστερμαν. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια, αγαπητοί συνάδελφοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Ιούνιο του 2013 διεξήχθη μια συζήτηση στην Σλοβενία όσον αφορά τις συστάσεις που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε και εμείς να συμμετέχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο στην φάση αυτή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η Επιτροπή που συνεδρίασε στη Σλοβενία αποφάσισε ότι οι συστάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι οι κατάλληλες. Θεώρησε ότι είναι ευεργετικέ για τη χώρα και ότι προσφέρουν τη δυνατότητα ανάληψης δράσης για την κυβέρνησή μας και ότι δεν αφορούν μόνο τη μεταρρύθμιση του συστήματος ταξιοδότησης της χώρας μου. Δεν είναι δυνατό αυτή τη στιγμή να έχουμε μια σφαιρική εικόνα όλων των κρατών μελών. Σίγουρα λοιπόν πιστεύω ότι οι συστάσεις αυτές πρέπει να είναι ειδικές αναχώρα. Οι δικές μας συστάσεις τουλάχιστον ήταν καλά προετοιμασμένες και στη δική μας την περίπτωση είχαν να κάνουν κυρίως με τις δημόσιες δαπάνες της χώρας μου με τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, με τη διασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης και επικεντρώνταν επίσης σε ορισμένους κλάδους της οικονομίας. Πρέπει επίσης να ασχοληθούμε περισσότερο και με μεταρρυθμίσεις στον τραπεζικό τομέα. Ο στόχος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είναι ο συντονισμός των εθνικών οικονομικών πολιτικών και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θεωρώ ότι θα ήταν ιδιαίτερα θετικό αν όλα τα κράτη-μέλη μπορούσαν όντως να συνεργαστούν όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση, ιδίω στα πλαίσια της Ευρωζώνης. Νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στην ε, αλληλεξάρτηση των οικονομιών μας και στις επιπτώσεις που αυτό ουσιαστικά προκαλεί. Ευχαριστούμε κυρία Όστερμαν. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Μπέρες, η πρόεδρος Επιτροπής Απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Euh, euh, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι πάρα πολύ σημαντική η δυνατότητα αυτή που έχουμε για να συνομιλούμε μαζί σας, αγαπητοί συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ακούσαμε ότι δεν αρκεί μια μισή ώρα, αλλά ξέρετε ότι ο διάλογος αυτός αποτελεί απλώς ένα τμήμα σε μια ολόκληρη σειρά διαλόγων που προβλέπονται στα πλαίσια του άρθρου 11 και στα πλαίσια του Fiscal Compact και μας επιτρέπει τελικά να συζητάμε πάρα πολύ συχνά και στο Βίλνιους τον επόμενο μήνα προφανώς. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να επιμείνω σε τρεις πτυχές. Πρώτον, για μας τους βουλευτές, είτε συμμετέχουμε στο εθνικό είτε στο ευρωπαϊκό κοινοβουλευτικό επίπεδο, οφείλουμε να πάρουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Συμβούλιο τελικά μια καλύτερη οριοθέτηση της όλη διαδικασίας, δηλαδή η εφετηρία των συστάσεων αυτών για χώρα να πρέπει να είναι προσαν... προσαντολισμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στη συνέχεια στα πλαίσια των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να μπορούμε τελικά να διαμορφώνουμε καλύτερα τις συστάσεις αυτές που γίνονται. Δεν γίνεται όμως κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη διάρθρωση ανάμεσα στην ετήσια επισκόπηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των συστάσεων αυτών. Να δούμε τελικά πώς μπορούμε στα πλαίσια της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης να διαμορφώνουμε καλύτερα τις ειδικές αναχώρα συστάσεις. Δεύτερη τώρα παρατήρηση. Πιστεύω ότι το Συμβούλιο στην, στα πλαίσια της προσέγγισής του αστικά υποτιμά τις πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει στρατηγική σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος ως προς τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Θεωρώ ότι υπάρχει μια αιμονή, για παράδειγμα, όσον αφορά να λαμβάνει την υπόψη το εργασιακό κόστος ως στοιχείο βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας σε μια χώρα, χωρίς να λαμβάνει την υπόψη ότι αυτό πραγματικά πειράζει πάρα πολύ τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό πραγματικά αγνοείται ή υποτιμάται στην καλύτερη περίπτωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό αποτελεί σημαντικό μέλημα για μας. Τελευταία τώρα παρατήρηση. Όσον αφορά το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο εξελίσσονται οι εθνικές μας οικονομίες, Προφανώς συμμερίζομαι και εγώ την άποψη ότι αν δεν έχουμε κοινωνικούς δείκτες και όσο δεν έχουμε κοινωνικούς δείκτες για να δούμε ποιες είναι οι μακροοικονομικές ανισορροπίες, τότε θα έχουμε μία προσέγγιση η οποία θα είναι μονομερής και η προσέγγιση αυτή δεν θα είναι καθόλου λογική και σωστά αιτιολογημένη από κοινωνική τουλάχιστον πλευρά. Είτε μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε μιλάμε ειδικότερα για την Ευρωζώνη. Τέλος, στην όλη αυτή γενικότερη προσέγγιση πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε κατά νου τη σημασία των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που λαμβάνουν χώρα και ιδίω την εφαρμογή της Τραπεζικής Ένωσης πραγματικά θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο για την ανάκαμψη των εθνικών και ευρωπαϊκών επενδύσεων σε πολλά κράτη-μέλη. Αυτή είναι η παρέμβασή μου. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε κυρία Μπερές. Το λόγο έχει η κυρία από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια για το εξαιρετικό της έργο. Ευχαριστώ και τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων που βρίσκονται εδώ για να κάνουμε αυτή την κοινή συζήτηση. Πιστεύω ότι είναι πολύ χρήσιμο και ωφέλιμο να ακούμε διάφορες απόψεις, διάφορες πτυχές διάφορες όψεις του ίδιου νομίσματος να βλέπουμε. Να κάνω ένα πρώτο σχόλιο σε ό,τι αφορά την χρονική συγκυρία και κατά δεύτερον ένα σχόλιο σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο των συστάσεων και το περιεχόμενο του εξαμήνου. Ως προς την χρονική συγκυρία θα ήθελα παρακαλώ να επιστήσω την προσοχή της κυρίας Φερέιρα στο ότι θα άξιζε τον κόμπο να δούμε πώς θα μπορέσουμε να συνάδουν, αν θέλετε, τα εθνικά, οι εθνικοί προπολογισμοί με το ευρωπαϊκό αυτό εξάμεινο. Γιατί είναι σημαντική αυτή η πτυχή. Σε ό,τι αφορά τώρα το περιεχόμενο και την χρησιμότητα του εξαμήνου, να λάβουμε υπόψη τα στοιχεία τα οποία ενδεχομένως να είναι χρήσιμα σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Κατά πόσον τα στοιχεία αυτά όντως επιφέρουν μια προστιθέμενη αξία. Κάθε χρόνο γίνονται οι σχετικές εκθέσεις οι οποίες και δίνουν και δείχνουν μια συνέχεια που υπάρχει. Συμφωνώ με πολλά από αυτά που ακούστηκαν από τα Εθνικά Κοινοβούλια ότι οι εκθέσεις αυτές για παράδειγμα αναφέρονται στο παρελθόν, το οποίο από μόνο του μπορεί να μην είναι πρόβλημα, αλλά θα πρέπει να υπάρχει κάποια πρόοδος, θα πρέπει να περιέχουν συστάσεις για το μέλλον. Να υπάρχει μια προοπτική μελλοντική δηλαδή. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει και τις συστάσεις αυτές χώρα λες και είναι κάτι το τελώς παγιωμένο που δεν τροποποιείται σε καμία περίπτωση. Αυτό θα ήταν σημαντικό να αλλάξει πάντα με απότερο στόχο να υπάρχει σωστός προϋπολογισμός, να προαχθεί η οικονομική ανάπτυξη, να προλάβουμε ενδεχομένως μακροοικονομικές ανισορροπίες. Προς αυτό το σκοπό όμως θα πρέπει να είναι παρόμοιες και οι μεθοδολογίες μας και ο τρόπος εξέτασης. Ο τεράστιος όγκος λοιπόν της εργασίας μας θα πρέπει να έχει καρπούς, να αποφέρει καρπούς. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε κυρία Γκαλπέλ. Τελευταίο τώρα ο είναι η συνάδελφος από την Κροατία, κυρία Μάντεριτς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την εισηγητριά μας για την πολύ καλή της έκθεση πολύ μεστή και λεπτομεριακή και θα ήθελα να χαιρετήσω και τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Αυτό που θα ήθελα να πω ότι ε, μία από τις προκλήσεις για την επιτυχή οικονομική πολιτική είναι ο συντονισμός των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών και ο μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου συμβάλλει στο συντονισμό των δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών μελών και με τον τρόπο αυτό βοηθά και στην ευθυγράμμιση, ε, την καλύτερη εναρμόνιση με την νομισματική πολιτική. Καλό θα ήταν να έχουμε μια κοινή πορεία στις δημοσιονομικές πολιτικές ε, και φυσικά να εφαρμόσουμε και τις κατάλληλες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Όλα τα κράτη-μέλη ουσιαστικά εστιάζονται στην υλοποίηση των στόχων που έχουν ε, εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το 2020. Και οι συστάσεις που είναι ειδικέ για κάθε χώρα είναι σημαντικές και κατά κάποιο τρόπο έχουν και έναν οριζόντιο χαρακτήρα γιατί με την ε, ανάλυση των συστάσεων αναχώρα μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι πολλές συστάσεις επαναλαμβάνονται. Ε, για παράδειγμα, η βελτίωση της δημόσιας διοίκησης, η, αναθεώρη, η ε, αναδιάρθρωση της αγοράς εργασίας, η αναδιάρθρωση του συνταξιοδοτικού συστήματος, η ενίσχυση της ε, αγοράς υπηρεσιών, η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η μείωση της ανεργίας, ιδιαίτερα της ανεργίας των νέων. Πρόκειται για συστάσεις που είναι κοινέ, είναι τομεί ε, και κοινή στόχη όλων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα η προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είναι ακριβώς η ανταλλαγή πληροφοριών ε, για να δούμε πώς ε, οι διάφορες χώρες εφαρμόζουν στην πράξη αυτά τα μέτρα. Και είναι χρήσιμη αυτή η ανταλλαγή απόψεων για να διαπιστώσουμε ποια είναι η εμπειρία της κάθε χώρας, για να διδαχθούμε από τις εμπειρίες αυτές και να αποφύγουμε ε, τα λάθη και από κοινού να συνεργαστούμε και να αντιμετωπίσουμε με τον πιο αποτελεσματικό και τον πιο γρήγορο τρόπο την κρίση. Ευχαριστώ. Muchas gracias, señora ευχαριστούμε κυρία Μάλετιτς. Ολοκληρώνονται εδώ οι παρεμβάσεις ε, των συναδέλφων ε, από τις ε, Εθνικές Βουλές και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ξαναδώσω το λόγο στην εισηγήτριά μας, την κυρία Φερέρα. Και πριν από αυτό θα ήθελα να πω ότι αν κάτι φάνηκε στη συζήτηση είναι ότι συμφωνούμε ότι οι εθνικές πολιτικές δεν είναι μόνο εθνικό ζήτημα, αλλά έχουν και μια ευρωπαϊκή διάσταση και οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε μια χώρα μέλος, ιδιαίτερα αν αυτή συμμετέχει στην Ευρωζώνη, έχουν άμεσα αποτελέσματα και αντίκτυπο και στα υπόλοιπα κράτη της Ευρωζώνης. Η κυρία Μπέρες μίλησε για το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και ο κύριος Έπινγκ εξέφρασε την ανησυχία του και το ενδιαφέρον του για την κατάσταση στην Ισπανία είναι φυσιολογικό η κατάσταση σε μια χώρα να ενδιαφέρει και τις υπόλοιπες ε, χώρες μέλη. Και φυσικά αυτά που συμβαίνουν στις, ε, στις κάτω χώρες ε, ενδιαφέρουν και απασχολούν και τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Όπως είπε ο κύριος Τρισέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουμε ένα κοινό πεπρωμένο. Η μοίρα μας είναι κοινή και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε με τη διαπίστωση αυτή. Χωρίς άλλη καθυστέρηση θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή σας και τις παρεμβάσεις σας και να δώσω και πάλι το λόγο στην εισηγητριά μας, την κυρία Φερέιρα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επαναλάβω τις θερμές μου ευχαριστίες για την πολύ ποιοτική συζήτηση. Ήταν πολύ επικοδομητικές οι παρεμβάσεις και πολύ χρήσιμες. Ε, περίτρανη απόδειξη ότι αυτή ε, η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου επιδέχεται με βελτιώσεων, αλλά σίγουρα αξίζει και είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Πολλοί συνάδελφοι μίλησαν ε, για τα θέματα αυτά. Δεν πρόκειται να αναφερθώ στον καθένα χωριστά, αλλά σημείωσα ε, τις παρατηρήσεις και θα προσπαθήσω στο μέτρο του δυνατού να τις συμπεριλάβω στο κείμενο που θα διαμορφώσω με τους σκιώδεις ηγητές, οι περισσότεροι από τους οποίους έλαβαν μέρος και στη συζήτηση. Θα προσπαθήσω λοιπόν να αντανακλώνετε και τα σχόλιά σας στην έκθεσή μου. Πολλοί αναφερθήκατε στην συγκεκριμένη συγκυρία και όπως θα διαπιστώσατε εγώ είμαι κάπως ε, μετριοπαθής. Εγώ δεν πιστεύω ούτε ότι έχουμε επιλύσει την κρίση, ούτε ότι έχουμε εξηγιάνει τα οικονομικά μας. Πιστεύω ότι θα πρέπει αυτά τα θετικά μηνύματα, αυτές τις θετικές ενδείξεις που ε, διαφαίνονται να μην ε, περιοριστούν εδώ και να αναπτυχθούν περαιτέρω. Ο κύριος Κοζές είπε ότι θα πρέπει να αξιολογήσουμε ε, αυτά που έχουν γίνει μέχρι στιγμής και μερικέ φορέ έχουμε την εντύπωση ότι τίποτα δεν έχει συμβεί. Όχι, όπω είπατε και εσεί ο ίδιος, αν δεν είχε γίνει τίποτα, ε, η Ελλάδα κατά πάσα πιθανότητα θα ήταν εκτό ευρώ και το ευρώ ίσω να μην υπήρχε πια. Όμω αντίθετα, πολλά έγιναν. Και η ανάλυση αυτή μα ενδιαφέρει για να δούμε αν αυτά που κάναμε, γιατί ε, κάναμε αρκετά, αν ε, αυτά που κάναμε όμω ήταν όλα σωστά. Ή αν υπάρχει περιθώριο να διορθώσουμε μερικά από τα πράγματα που κάναμε. Γιατί βλέποντα και την αντίδραση άλλων εταίρων μας ε, στην κρίση, όπω των Ηνωμένων Πολιτειών, διαπιστώνουμε ότι έχουμε αρκετά να διδαχτούμε από τους υπόλοιπου εταίρου. γιατί δεν είμαστε εμεί ε, ούτε τέλειοι ούτε αλάθετοι και οι στρατηγικές μας ε, έχουν και αυτές κάποια λάθη και καλώς ε, θα, καλό θα ήταν να τα διορθώσουμε και να χρησιμοποιήσουμε αυτή την κρίση για να ενισχύσουμε τη θέση μας. Δηλαδή να γεφυρώσουμε τα κενά που υπάρχουν ακόμη στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα και να χρησιμοποιήσουμε τους υφιστάμενους μηχανισμούς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ήταν ε, σημαντικές κάποιες ε, παρεμβάσεις που έγιναν για τα περιθώρια πρόοδου που έχουμε για παράδειγμα, η Τραπεζική Ένωση σίγουρα είναι ένα τομέα στον οποίο θα σημειώσουμε πρόοδο και αυτή τη στιγμή ο κύριος Λανσουέλα μίλησε για κάποια σταθεροποίηση και είναι σημαντικό που έχουν δημιουργηθεί τα OMTs από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και έχουν δημιουργηθεί διακυβερνητικοί μηχανισμοί όπως είναι ο μηχανισμός σταθερότητας. Είναι σημαντικά όλα αυτά τα στοιχεία και θα πρέπει να τα δούμε και υπομέσω και μακροπρόθεσμη προοπτική. Ούτε μπορούμε να υποβαθμίζουμε όλα αυτά που έγιναν όπως το blueprint της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή το κείμενο των τεσσάρων προέδρων. Γιατί με το κείμενο αυτό έχουμε ένα πιο μακρόπονο όραμα, μέσο και μακροπρόθεσμο και της Νομισματικής Ένωσης αλλά και της ε, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τους μηχανισμούς που έχουμε, όπως είναι αυτός του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και του συντονισμού των δημοσιονομικών πολιτικών. Γιατί έχουμε κάποια σημάδια ανάκαμψης, μεν, αλλά δυστυχώς η ανεργία εξακολουθεί να είναι σε ανυπόφορα επίπεδα. Επίσης έχουμε δημόσια χρέη σε πολύ ψηλά επίπεδα. Έχουμε φαινόμενα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού που είναι οξύτατα και σοβαρότητα. Οπότε από πολιτική άποψη θα πρέπει να ενισχύσουμε ή να αναζωογονήσουμε την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών στην Ευρώπη και στην ικανότητα της Ευρώπης να αντιμετωπίσει πολιτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Τώρα, στα πλαίσια του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών θα πρέπει όλα αυτά τα στοιχεία να τα λάβουμε υπόψη. Θεωρώ ότι μία αναδιατύπωση του μηχανισμού της Τρόικας ε, στα πλαίσια του έργου του διπλού πακέτου είναι πολύ σημαντική, όπως μας ε, είπε και ο κύριος Γκοζές. Είναι επίσης σημαντικό να διευκρινίσουμε όλους τους μηχανισμούς ε, για την ανταγωνιστικότητα και τη σύγκληση και της πρωτοβουλίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα CCI, που θα πρέπει να εφαρμοστούν γιατί θα, συνδράμουν τα κράτη-μέλη στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και θα συμβάλλουν ως κίνητρο και όχι μόνο ως κύρωση για να υλοποιηθούν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και επίσης θα πρέπει να εφαρμοστεί μια ελαστικότητα στους βαθμούς προσαρμογής. Θα δούμε τώρα πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ε, χρησιμοποιήσει την ελαστικότητα στο εξαπλό και το διπλό πακέτο στον προπολογισμό του 2014 για να ενισχύσει την επένδυση εν ώψη της στρατηγικής του 2020 και πώς θα συντονιστούν τα θέματα του δημοσίου χρέους στην νέα ομάδα που δημιουργήθηκε. Ε, Πολύ αναφέρθηκαν στην ποιότητα των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κυρία Γκάλ Πέλτς ε, μίλησε για το θέμα αυτό και μία άλλη ε, βουλευτής επίσης. Είναι σημαντικό να αξιολογήσουμε τις συστάσεις αυτές, όχι μόνο από άψη ποιότητας και βελτίωση της ποιότητάς τους, αλλά να κάνουμε αυτά που είπαν ο κύριος Λίντς, ο κύριος Καμπρίτο και πολλοί άλλοι βουλευτές, να εκδημοκρατήσουμε τη διαδικασία αυτή. Ο εκπρόσωπος της Γαλλικής Ιθνοσυνέλευσης επίσης το τόνισε. Θα πρέπει οι χώρες μέλη να ε, στενιστούν αυτές τις συστάσεις, να τις νιώσουν ως δικές τους και φυσικά να αξιολογήσουν τη ποιότητα αυτών των συστάσεων κάνοντας μία επανισορρόπηση μεταξύ της ανάγκης ε, του δημοκρατικού χαρακτήρα ε, κάθε χώρα και αναγνωρίζοντα ταυτόχρονα ότι οι χώρε πια δεν είναι ελεύθερε να ακολουθήσουν τι πολιτικέ του μόνε του, γιατί οτιδήποτε κάνουν και οτιδήποτε αποφασίζουν έχει αντίκτυπο στι υπόλοιπε χώρε. Θα πρέπει να γίνει με στη διοργάνωση λοιπόν αυτών των μηχανισμών συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Θα πρέπει να επεξεργαστούμε καλύτερα αυτό αυτούς τους μηχανισμούς συνεργασίας. Ο κύριος Λίντς μίλησε για, την αρχιτεκτονική της συμμετοχής. Είναι πολύ σημαντικό να το επεξεργαστούμε αυτό το θέμα και οι συστάσεις, ναι μεν είναι ε, της Επιτροπής και του Συμβουλίου, αλλά θα πρέπει να έχουν μια δημοκρατική νομιμοποίηση, θα πρέπει να έχουν το στίγμα της δημοκρατίας, ε, να λαμβάνουν την έγκριση των ε, ερετών είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν να ε, δώσουμε έμφαση σε αυτό το δημοκρατικό χαρακτήρα των συστάσεων. Επίσης, ε, τι γίνεται με τις πολιτικές εκτάκτου ανάγκες. Θα πρέπει και αυτές να τις λάβουμε απόψη, καθώς και την κοινωνική πτυχή, με σημαντικές πρωτοβουλίες τόνωσης ε, της απασχόλησης και ε, κοινωνικής αλληλεγγύης. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε διάσπαση κοινωνική εξαιτία των ευρωπαϊκών πολιτικών. Σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό και υπάρχει ανάγκη κατεπηγόντως ε, να ανασκομποθούμε και να δούμε και τους ε, ε, κοινωνικούς δείκτες αλλά και να προτείνουμε πρωτοβουλίες για την απασχόληση. Γιατί Καλές είναι οι πρωτοβουλίες ε, μέσω και μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξη, αλλά θα πρέπει να ξεχνούμε και την βραχυπρόθεσμη προοπτική. Και βραχυπρόθεσμα θα πρέπει να αναζωογονήσουμε την ευρωπαϊκή οικονομία με λογικό, στρατηγικό τρόπο, μέσω και μακροπρόθεσμα, αλλά και βράχυπρόθεσμα. Και η κυρία Μπέρες ε, και άλλοι συνάδελφοι το ανέφεραν. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η φάση, γιατί η σοβαρότητα της κρίσης που διανύσαμε και που διανύουμε τα τελευταία χρόνια μας ε, κατέσαν επιτακτική την ανάγκη να διορθώσουμε τα κενά που υπάρχουν, να τα καλύψουμε και ταυτόχρονα να επιτύχουμε μεγαλύτερη σύγκληση, να εντείνουμε τις προσπάθειες σύγκλησης και συντονισμού για βασικά θέματα οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Και τελικά ελπίζω ότι η έκθεσή μου θα αντικατοπτρίζει όλα αυτά τα μηνύματα που μας μετέφεραν τα Εθνικά Κοινοβούλια. Και από αυτή την άποψη θεωρώ ήταν πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η συνάντηση. Σας ευχαριστώ θερμά. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Φερέρα. Θα ήθελα να σας ανακοινώσω τώρα ότι η ψηφοφορία τη έκθεση της κυρίας Φερέιρα στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων θα γίνει στις 30 Σεπτεμβρίου ε, και η έκθεση θα περάσει την Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Θα ήθελα θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφου από τα Εθνικά Κοινοβούλια για τις παρεμβάσει του ε, και τα σχόλιά τους που θα συμπεριληφθούν και θα εμπλουτίσουν και το δικό μας έργο και να σας ε, υπενθυμίσω την επόμενη μας ε, κοινή συνάντηση που θα γίνει τον Ιανουάριο στα πλαίσια της διακοινοβουλευτικής ε, συνέλευσης για να κάνουμε την συζήτηση για την ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης, το Annual Growth Survey, που θα εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 15 Νοεμβρίου. Επόμενο σημείο της σα διάταξης είναι τα διάφορα. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει τίποτα για τα διάφορα. Οπότε το τελευταίο σημείο, αυτό που σας είπα, η επόμενη μας συνεδρίαση θα γίνει στη Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου, 3 με 6.30 και την Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου, 9 με 12.30 και 3 με 6.30. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας απόγευμα, ελίεται η συνεδρίαση.